Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Επίτροπο, στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Καλημέρα σε όλου του αξιότιμου συναδέλφου, άντρε και γυναίκε. Ξεκινάμε τη συζήτησή μα. Ξεκινάει η συνέδριαση. Πρώτο σημείο τη